Hey colleagues. We've got to carry on the votes now. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες μας. This is the draft report on the proposal. για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνηση επιβίβαση σηματέωση μεγάλη καθυστέρηση πτήση και τροποποίηση του κανονισμού υπαριθμών 2027-97. Έτοιμοι. 180. Υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, πέρας της ψηφοφορίας. Α, περιμένουμε το συνάδελφο να τοποθετεί στην κάρτα του. Εγκρίνεται ούτως ή άλλως, 25-11. 181 και 22 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για να πάρω μια ιδέα για τον αριθμό των ψήφων. άρχιε η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 24 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 182. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 και ήμικο 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι επόμενες δύο καταπίπτουν άρα πάμε στην 23 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 για τις έκτακτες ε, συνθήκες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν μου αρέσει η άποψη των αεροπορικών εταιρείων για αυτές τις ε, έκτακτες ε, συνθήκες. 199 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ψηφίσουμε τη 206 ηλεκτρονικός. Έναρξη παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι υπέρας. Απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 210 και 211 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 213 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στη 213 έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Γίτσες κύριε Χέρτσοκ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 και 221 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 222 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 223. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη, 27 και 29 της ΣΥΜΚΟ είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ε, της 232 νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά επειδή έχουμε πάθει, έχουμε αγγυλωθεί τα χέρια μας πάνω κάτω Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Πέρας της ψηφοφορία. εγκρίνεται. 233. Παρακαλώ, σηκώστε καλά τα χεράκια. Υπέρ. Υπέρ και λέω στους σοσιαλιστές κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Το δικό σας χέρι για του κυρίου Φρίγκου ήταν τα μόνα που σηκώθηκαν. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Λοιπόν, 31 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έλεγξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. πέρας. Εγκρίνεται. 29. 29. Υπέρ. Όχι, καταπίπτει, καταπίπτει. Συμβιβαστική 5. Ε, πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 239. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. ούτως ή άλλως απορρίπτεται. Μήπως μπορείτε να καθίσετε δίπλα στο Σπύρο, ίσως καλύτερα. Δεν το κατάλαβα. Ο κύριος Lightfoot δεν είναι εκεί. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως πάμε στην τροπολογία 31. Του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν 2.41. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ψηφίσουμε τη 241 το πρώτο της τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Άρα απορρίπτεται, άρα το δεύτερο τμήμα δεν έχει νόημα το ψηφίσουμε. 242 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 και 243 μαζί είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 244, 45 και 33 και 34 από ήμικο καταπίπτουν. 246 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 247 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται 248 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 260. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 260. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 34 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει, καταπίπτει. 261 ψηφίζουμε τώρα. 261 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 262-263 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικός έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Περάς. Απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά έναρξη ψηφοφορία. Everybody Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονικός έλεγχος της 267 έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πάλι σοπαλία, πάλι απορρίπτεται. 35 ε, με προφορική τροπολογία 2. Διαφωνεί κανεί Αν όχι, την ψηφίζουμε μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 269 είναι η επόμενη τροπολογία μας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχο της 269. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 288 καταπίπτει. 41 έχει αποσυρθεί. 287 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 293 είναι γλωσσική Ήμικο 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος της 295. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ισοπαλία. Απορρίπτεται 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μέχρι τη 299 καταπίπτουν. Οι 45 και 44 τσίμκο είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 331. Είστε εδώ? Ωραία. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 332 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 333 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 49 υπέρ. Κατά. Άποχες η ηλεκτρονικός έλεγχος της 49 της ΣΥΜΚΟ, ένδοξη πληροφορία. Ψηφίσατε όλοι. Περάς. Πάλι ισοπαλία, πάλι απορρίπτεται. 334 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 335 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 361 υπέρ κατά αποχές Μπορούμε να ελέγξουμε την 361. Έναρξη. Συμφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Γιατί κανείς δεν σήκωσε το χέρι. Λοιπόν, έναρξη ψηφοφορίας για την 53. Ψηφίσατε όλα, όλοι. Ε, είστε σίγουροι ότι ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας. Εγκρίνεται. στην 364. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 367 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 367. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 369 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 366 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες. Πάμε στην 372. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 373 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 374 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 385 τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61. Και σύμικο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 398 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 και 400 καταπιπτούν. Την 63 ψηφίζουμε. Τη ΣΥΜΚΟ ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. πορύπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 401 και 403 μαζί υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις δύο παρακαλώ. Έναξη ψηφοφορίας. 401 και 403 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το 410 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Ναι, ναι, απερίφθη. 411 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 64. Ψήφισαν όλοι. Ε, από τους Άλντε υπάρχει ένας παραπανίσιος. Διορθώστε το παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 412 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 του εισηγητού. Α, η 411 δεν εγκρίθηκε, επομένως Επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.13 ως προσθήκη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.15 υπέρ, κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την, ψηφο... για την τροπολογία 415 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 417. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4.18 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 4.18 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Συμβιβασμός 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 427, 27, 428, 429, 430, 68 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 431 καταπίπτει. Η τροπολογία 69 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. αποχέσε, Επαλήθευση παρακαλώ. Γιατί κανένας πια δεν ψηφίζει. Η τροπολογία 69 της ΙΜΚΟ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 70 της ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 70 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 432 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 439 Τροπολογία 439 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 440 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 της ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.45 υπέρ Τέσσερα σαράντα πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα σαράντα έξι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 21. Συμμαζέψτε το μυαλό σας, λέει ο πρόεδρος. Συμβιβασμός 21. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 451. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 452 ως προσθήκη. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 453 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 447 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 467 καταπίπτει. 463 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4,55 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, αλλά σας το λέω, εδώ αριστερά δεν ψηφίζει κανένας, δεν σηκώνει κανένας το χέρι του. Τροπολογία 76, μα βοηθήστε με λίγο, δεν μπορώ να είμαι medium να διαβάζω τις επιθυμίες σας χωρίς να σηκώνετε το χέρι σας. Σαΐντ, ε, αν δεις το χαρτί σου, το 76 δεν έχει μείον, έχει συν. Είναι η τροπολογία 76 του εισηγητού. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 76. Τροπολογία ΙΜΚΟ 76. Those in favor. Those Αυτό έχει μείον. Αποχές απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές 458 να την ελέγξουμε, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 459 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 460 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 461 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 78 υπέρ. Τι δεν τις βρίσκω. Εγκρίνονται. 464 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 466 466 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση 466. Ηλεκτρονική επαλήθευση 466. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε. Συμβιβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 483 ως προσθήκη υπέρ. 483 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα ενενήντα ένα με μια προφορική τροπολογία υπαριθμών τέσσερα. Υπάρχει κάποια αντίθετη γνώμη για την προφορική τροπολογία, όχι, επομένως ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 492 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 494 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 495 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 496 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 497 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 88 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 500 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 500, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη η τροπολογία 500. Τροπολογία 82 ΙΜΚΟ, αυτή καταπίπτει ούτως ή άλλως, επομένως 4,99. Όχι, 4,98. Καταπίπτει και η 4,98. Και η 4,99 καταπίπτει. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 501 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 501 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 502 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 503 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 504 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 505 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 505, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας, αποτέλεσμα απόρριψη. 506 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 469 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 508 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 509 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 511 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 513 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 507 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 512 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.16 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5.18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5.19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Συμβιβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. How many more Πόσες σελίδες ψηφοφορίας έχουμε ακόμα? IMCO as an addition, those... Τροπολογία IMCO 86 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. ΙΜΚΟ 86 ως προσθήκη. Μόνο πέντε ψηφίσανε προηγουμένως. Για να δούμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ε, ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 524. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 87 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 5.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.26 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 529 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Οι 5.30 και οι 5.31 είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 27, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 541 και 542 είναι ταυτόσημες, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4, ε, συγγνώμη, 549 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν ΙΜΚΟ 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 98 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. πρέπει να ψηφίσουμε και την τροπολογία ΙΜΚΟ 92 που την ξεχάσαμε υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 5.55 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.54 καταπίπτει. Ε, το ίδιο και το δεύτερο τμήμα καλύπτεται από την τροπολογία 99 όπως γράφει το χαρτί μου. Άρα πηγαίνουμε στην 99 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 556 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 558 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 94 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβασμός 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μ' αρέσει αυτός ο συμβιβασμός, είναι χορταστικός. Τροπολογία 107 στα αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 107, τη βρήκατε όλοι. Πολύ ωραία ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία 108, κατά τμήματα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, τώρα μαζί με τις λέξεις που είχαμε απορρίψει πριν, αποκλείσει πριν, υπέρ, υπέρ στην πλήρη διατύπωση, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αυτή ήταν η τροπολογία 108 που μόλις ψηφίσαμε. Ενεκρίθη λοιπόν με το κείμενο indirectly κλπ. Τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 112 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 112 άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 115. Υπέρ. <coughs> Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 1. Καταπίπτει ήμκο 1. Α, τώρα σαν προστίκη. Υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 116 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για το 116. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τροπολογία 114 είναι γλωσσική, 117 είναι η επόμενη, υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 119 υπέρ κατά Αποχέσε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 119 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 118 υπέρ κατά αποχέσε. απερίφθη. 120 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 120 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Κουράγιο, σε λίγο τελειώνουμε. And it's rejected. Απερίφθη. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές. Παρακαλώ να ελέγξουμε τροπολογία 123 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη. 124 υπέρ Α, καταπίπτει, ναι, ναι, καταπίπτει, καταπίπτει. Τροπολογία 5 του εισηγητού, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 2 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Ήμκο 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 4 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφολική τροπολογία 7 του εισηγητού Συμφωνείτε με την ε, κατάσταση προφορικής τροπολογίας. Ναι, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, πού πρέπει να πάμε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 9 καταπίπτει. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 136 καταπίπτει, 137 ως προσθήκη. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 138, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται η τροπολογία 138. 141-142 είναι ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ήμκο 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η 145, 146 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. Προφορική τροπολογία 5, υπάρχει αντίρρηση, όχι, επομένως ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. Ίμκο 15 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίμκο 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 153 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τροπολογία 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. ΙΜΚΟ 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 16 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 157 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 καταπίπτει. Όχι, όχι, είναι, συγγνώμη, ε, θα την ψηφίσουμε ως προσθήκη. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 καταπίπτει. Ε, λόγω της τροπολογίας 158 φτάνουμε στην 160 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 161 είναι μέρος του συμβιβασμού, επομένως 162 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 163 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 164 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 165 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη, τροπολογίες 166 και 167 είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Τροπολογία 168 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 169 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 ΙΜΚΟ ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 171 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία ΙΜΚΟ 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 172 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία ΙΜΚΟ 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 173 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 174 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 177 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχέσε απερίφθη. Τελική ε, ψηφοφορία άρχεται, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 37 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Το ε, νομοθετικό ψήφισμα, νομοθετικό ψήφισμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 37 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή, επομένως εγκρίνεται και το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου και συγχαίρουμε τον συνάδελφο Ζόρζ Μπαχ. Ωραία, επόμενο θέμα στη σε διάταξη. Ησυχία σας παρακαλώ. ή αφορά τη Διεθνή Σύμβαση το Ρεμολίνος του 1970 για την ασφάλεια των αλλιευτικών σκαφών. Πρόκειται για μια ε, έκθεση του κυρίου Κούν να πω στους συναδέλφους εάν θέλουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να την εγκαταλείψουν ησύχω. Ο κύριος Κούν. Ε, um Πρόκειται για μια συμφωνία του 2012 από το Cape Town Συμφωνία του Cape Town λοιπόν. Το 1977, μια διεθνή συμφωνία, και αυτό είναι το υπόβαθρο, του Τωρεμολίνος συγκεκριμένα συνήφθη μια διεθνή συμφωνία που αφορά την ασφάλεια των αλληλευτικών σκαφών. Το 1993 το πρωτόκολλο προσαρτήθη στην συμφωνία του 1977, προσαρμόστηκε συνθήκες έγινε επεξεργασία των σημαντικότερων κεφαλαίων, συμπεριλήφθηξαν περιφερειακή διάσταση και έτσι από 24 μέτρα και πάνω τα λευτικά σκάφη καλύπτονται από αυτήν τη συμφωνία του Τωρεμολίνος. Πλην όμως, πλην όμως το πρωτόκολλο αυτό δεν ε, τέθη ποτέ σε ισχύ γιατί δεν, έγιναν, δεν υπήρξε επαρκής αριθμός κυρώσεων από τα κράτη-μέλη. Και έτσι στο Cape Town μια διπλωματική διάσκεψη που ε, συγκάλεσε η Διεθνής Ναυτιλία, ε, Οργάνωση Ναυτιλίας είχε σαν στόχο να εξασφαλίσει περισσότερη υποστήριξη για το πρωτόκολλο και γενικά για την ασφάλεια των σκαφών, ανεξαρτήτως του αν είναι αλλιευτικά, επιβατικά και Πρόκειται δηλαδή για πρόσθετες συνθήκες ασφαλείας πέραν αυτών που απαιτούνται για τα αλλιευτικά σκάφη, αλλά και ιδιαίτερως για αυτά που έχουν ιδιαίτερες συνθήκες, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η συμφωνία λοιπόν του 2012 για την υλοποίηση ε, για την εφαρμογή των ε, διατάξεων του 1993 για την ασφάλεια των ε, αλληλευτικών σκαφών έτσι πλησιάζει στην πραγματοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 97-70 ε, για την εναρμονισμένη νομοθεσία τη σχετική με τα σκάφη από 24 μέτρα και άνω ε, εφαρμόζει τις διατάξεις αυτές από το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν είναι, και αυτή είναι η δυσκολία, άμεσα συμβαλόμενο μέρος σε αυτή τη συμφωνία με τη Διεθνή Οργάνωση Ναυτιλίας. Τα κράτη-μέλη, το καθένα χωριστά δηλαδή, πρέπει να υπογράψουν. Και μόνο, βέβαια, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να το πράξουν αυτό τα κράτη-μέλη. Εφόσον υπάρξει σχετική παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο ή με σχετική επαφή του Κοινοβουλίου. Είναι διαρθρωμένη λοιπόν έτσι η συμφωνία, ώστε προβλέπει 12 μήνες μετά τη θέση ισχύ της, να ε, να αρχίζει να είναι δεσμευτική. Χρειάζεται όμως τουλάχιστον 20 κράτη να κυρώσουν. Ιδάλλως δεν έχει και κανένα νόημα και αφορά πολύ λίγα ε, αλληλευτικά σκάφη, 3.600 συγκεκριμένα. Τώρα λοιπόν διευκολύνεται αυτός ο όρος με 15 κράτη πλέον και 14.000 αλληλευτικά σκάφη. Μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου λοιπόν του 2014 είναι ανοιχτή, από τις 11 Φεβρουαρίου του 2013 στις 10 Φεβρουαρίου του 2014 ανοιχτή για υπογραφή στη Εθνή Ναυτιλιακή Οργάνωση, η Συμφωνία. Και όπως είπαμε τώρα τα κράτη-μέλη πρέπει ή μπορούν καλύτερα να δηλώσουν είτε με κύρωση είτε με προσχώρηση, την, προσχώρηση στο πεδίο εφαρμογής την ε, συμφωνία αυτή. Υπάρχουν ε, για να διευκολυνθεί η αποδεξιμότητα της συμφωνίας ε, πιο ελαστικές διατάξεις για τους εξοπλισμούς, για τις ραδιοεπικοινωνίες, για τα σωστικά μέσα. Άλλο ούτως ή άλλως πάντα ισχύουν οι διεθνείς διατάξεις. Και μια άλλη δυνατότητα για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής με πρόσθετες δηλώσεις μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να διαρθρώσουμε περισσότερο τις ε, θέσεις μας, αλλά πάντως το βασικό να γίνει η εφαρμογή. Οι επιθεωρήσεις των προϊόντων που θα προκύψουν ε, θα γίνεται από την αρμόδια διεθνή αρχή ασφαλείας, θα γίνουν οι προσαρμογές, οι τροποποιήσεις που χρειάζονται και εποπτεία επιθεωρήσεις εφόσον βεβαίως ε, γίνουν όλες οι προσαρμογές εγκαίρως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συμφωνία γιατί στον τομέα αυτών ε, των αλληλευτικών σκαφών έχουμε πολλά ατυχήματα, είτε άμεσα συνδεδεμένα με την αλληλεία και την ε, κατεργασία του αλληλεύματος στο σκάφος και βεβαίως αυτό σημαίνει πολλές ανθρώπινες ζωές 24.000 άνθρωποι χάνονται κάθε χρόνο ή υπάρχουν ατυχήματα σχετικά και βέβαια και στις διεθνείς μεταφορές μπορούμε να εξασφαλίσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ή μη τι άλλο περιορισμό των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζει εφόσον περισσότερα κράτη-μέλη προσχωρήσουν στην αλληλευτική αυτή συμφωνία, εφόσον εξασφαλίσουμε την προσχώρηση, γιατί έτσι αλλάζουν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα αλληλευτικά σκάφη με το που θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Αυτό που μπορώ να πω λοιπόν εγώ από πλευρά μου είναι οπωσδήποτε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε, άλλωστε άλλη δυνατότητα γιατί πρόκειται για εκτελεστική πράξη δεν έχουμε. Thank you very much. it is a consent procedure. Άρα πρόκειται για διαδικασία σύμφωνη γνώμη. Είτε ναι είτε όχι λέμε, δεν έχουμε να αλλάξουμε τίποτα. Κυρία είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μας το εξηγήσατε. Είναι πάρα πολύ παράλογο το ότι δεν μπόρεσε τόσα χρόνια να τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία. 15 κράτη μάλιστα, με 14.000 σκάφη ήταν η αρχική ε, πρόθεση, τώρα γίνανε 22 με 3.400 κάτι, δηλαδή έχουμε πιο πολλά κράτη, αυτό είναι ίσως θετικό, με λιγότερο όμως σκάφη. Και άρα ίσως είναι και πιο εύκολο να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη προς των κρατών. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύσει αυτή η συμφωνία ε, όπως και να έχει με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τα ε, σκάφη με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όπως και για τα άλλα. Και κάτι άλλο, τα τώρα σκάφη τα οποία ε, έχουν ελευτικές δραστηριότητες στα νερά μας, στα υδατά μας, ε, είναι μικρότερα, έχουν μήκος μικρότερο από 24 μέτρων. Και άρα όπως υπόθηκε και νωρίτερα μπορεί να είναι αυτή η συμφωνία κατάλληλη και για τα πιο μικρά σκάφη. Πάντως πιστεύω ότι πρέπει να πούμε το ναι, γιατί έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά τα ε, τις συνθήκες ασφαλείας για τα λευτικά σκάφη ύστερα από 20 τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αν όχι... Έχουμε εδώ την εκπρόσωπο της Επιτροπής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και το Κοινοβούλιο για την ε, ταχύτατη ε, συζήτηση και διαπραγμάτευση του θέματος αυτού. Τον Οκτώβριο του 2012 ήρθε αυτή. Χαίρετε, εδώ είμαι. Ε, ήρθε η πρόταση, η πρόταση της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2013. Είχαν τα κράτη-μέλη εκδηλώσει κάποια ανάγκη για περισσότερο χρόνο, είχαν ζητήσει περισσότερο χρόνο περιοκειμένου να εξετάσουν τις, ε, τα κείμενα και τις επεξηγήσεις που τα συνόδευαν. εδώ προκειμένου να μην γίνει χρήση των εξαιρέσεων οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία και που δεν έχει εφαρμοστεί από το 1997. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται λοιπόν να δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν χρήση των εξαιρέσεων, θα δηλώνουν στη Διεθνή Οργανώση Ναυτιλίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούμε εμείς από την Επιτροπή, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν δώσει τώρα τη συνένωσή του και έτσι οι συμφωνίες στο Ρεμολίνος και Cape Town ε, τεθούν σε ισχύ, μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε σε διεθνές επίπεδο την ε, διατήρηση των όρων, την εφαρμογή των όρων ουσιαστικά αυτή τη ευρωπαϊκή τελικά οδηγία και νομίζω ότι θα έχουμε εξυπηρετήσει στα μάλα τον κλάδο των αλληλευτικών σκαφών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, Προθεσμία για τι τροπολογίε 19 Δεκεμβρίου. Η μόνη τροπολογία, υπενθυμίζω, είναι αυτή που προτείνει απόρριψη. 19 Δεκεμβρίου προθεσμία λοιπόν, 21 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Κύριε Κούν, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έχουμε τα δύο μέτρα για τα πλοία ιστορική ναυσιπλοεία, ο κυρία Βόρτσμαν Κόρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Γκρός. Ε, λαμβάνει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφο ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, αλλά μου έχει δώσει τι προτάσει τη. Έχουμε λοιπόν τι εκθέσει για, ε, για τα πλοία εσωτερική ναυτιλία. Ξέρετε ότι, θα, ότι υπήρχε ένα ταμείο το οποίο είχε στη θέσή του 35 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν, αν δεν κάνω λάθο, με περιορισμένη όμω αξιοποίηση εν τέλει και απορρόφηση κονδυλίων. Και έτσι έρχεται μια πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή του ταμείου αυτού, έτσι ώστε να καλύψει και την ε, ε, επιμελητία. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συγκέντρια συγκεκριμένα. Και υπογραμμίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε ε, πιστοί στον όρο ότι δεν πρέπει να ενισχύεται ο στόλος, να μην γυρίζουμε δηλαδή στο παρελθόν. Γιατί αυτό το ταμείο έχει και σαν στόχο την ε, αντικατάσταση των ε, παλαιών ε, από νεότερα σκάφη, αλλά όχι η αύξηση του δυναμικού, του ελευτικού δυναμικού. χαιρετίζει λοιπόν η κυρία Βόρτσμαν Κόλ την συνεργασία που αναπτύχθηκε στο χώρο της ε, εσωτερικής ναυσιπλοείας και των μεταφορών της πλωτής οδού. Ε, πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την επίτευξη των τεχνολογικών προδιαγραφών, τεχνικών προδιαγραφών. Έχει κάνει ίδια κάποιες τροπολογίες γιατί δεν είναι 100% σίγουροι ότι είναι επαρκείς οι προτάσεις, όχι γιατί πρέπει να γίνει προσαρμογή των παραρτημάτων, αλλά γιατί θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η αρχή της συνεργασίας. Και τρίτον χαιρετίζει και την πρόταση να, κάτι κάνουμε κι εμείς καλό και με του συντονιστέ, κύριε Πρόεδρε και που αποφασίσαμε χθε στη διάσκεψη των συντονιστών την προφορική ερώτηση για την ε, ε, επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης ε, γιατί και πολύ λίγο διάστημα πριν από τις εκλογές καλό είναι να ακούγονται αυτές οι προτάσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια έννοια όχι απλώς θεωρητική αλλά κάτι το πολύ απτό, κάτι με σάρκα και ωστά. και πρέπει να το δούμε. Ευχαριστεί λοιπόν η συγγετρία του συναδέλφους για τις παρατηρήσεις πολύ ευγενικέ και υποθετικές και θα συνεχίσει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Σαρτού, Αρτού. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε πρόεδρε, συμφωνώ με τις εισηγήτριες ε, και στην Επιτροπή και της Επιτροπής Απασχόλησης ε, και της δικής μας Επιτροπής ως προς το, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του Ταμείου, του κανονισμού δηλαδή συγκεκριμένα όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ταμείο αυτό, το αποθεματικό των 35 εκατομμυρίων ευρώ ε, πρέπει βεβαίως να αξιοποιείται προς όφελος των δικαιούχων. Σε αυτό συμφωνούμε και για τους επιχειρηματίες βεβαίως όπως και για τους εργαζομένους θα πρέπει να διατεθεί κατά ισότιμο τρόπο η υποστήριξη από το Ταμείο αυτό. Από την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης έχουμε μια αναφορά στην ε, πρώιμη σταξιοδότηση, στις ε, δεξιότητες, στην επίσημη, η τυπική μάλλον κατάρτιση ως προϋποθέσεις για τη διάθεση των κονδυλίων. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπουμε με ικανοποίηση ότι υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η στόχευση της εναρμόνισης των προδιαγραφών και της ενίσχυσης ε, στη διεθνή συνεργασία. Η εναρμόνιση θα πρέπει να γίνει σε τομεακό επίπεδο, σε αυτό συμφωνώ με την εισηγήτρια. Άλλωστε το συζητήσαμε, είπαμε δηλαδή ότι η Κεντρική Επιτροπή Ρήνου ε, και η αρμόδια υποεπιτροπή της θα πρέπει να δώσουν πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Επίσης, ως Κοινοβούλιο πιστεύουμε και επιμένουμε ότι δεν πρέπει να τροποποιηθούν τα τεχνικά παραρτήματα, αλλά πρέπει απλώς να εξυπηρετηθεί ο στόχος της δημιουργίας ενός πλαισίου ε, για, τις τεχνικές, για τη λειτουργία αυτών των τεχνικών προδιαγραφών και επίσης ε, συμφωνούμε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τις ε, αρμοδιότητες για την προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε, άλλους αντίστοιχους, σε άλλα αντίστοιχα νομοθετήματα. Βεβαίω ε, είναι πολύ πιο οικολογικός αυτός ο τρόπος μεταφορών, οι πλωτές μεταφορές και πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξουμε την ακόμη, περισσότερο, την ακόμη πιο οικολογική διαμόρφωσή του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σμάισνερ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα πείτε βέβαια κύριε Γκρό την κυρία Βόρτσμαν Κόρα που δεν είναι εδώ πως την ευχαριστώ. Είχαμε ε, πολύ καλή συνεργασία με τις ορσκιώδης γιατί Πετρή και εγώ. Ε, βεβαίως μπορούμε να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά, να αποφύγουμε την επικάλυψη εργασιών και νομίζω ότι εάν ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την κατάρτιση μπορούμε πολλά πράγματα να κερδίσουμε. Αυτό ως πρώτη παρατήρηση και μια και υπάρχει και ένα δεύτερο τμήμα αυτά τα 35 εκατομμύρια ευρώ είναι παράλογο το ότι δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί γιατί δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις και δεν υπήρχε δυνατότητα να απορροφηθούν. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει το χέτερο δηλατός. αυτό συμφωνούμε απολύτως, πρέπει να αναπτυχθεί ο τομέας, πρέπει να σπρώξουμε τις μεταφορές από τους δρόμους στις πλωτές οδούς και γι' αυτό το στόχο θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τα μέσα που θα μας βοηθήσουν. Είχαμε ένα τριμερή διάλογο για τις εναλλακτικέ υποδομές, μάλλον τις υποδομές για τις εναλλακτικέ μορφές ενέργειας, όπου και οι πλωτές οδοί, γενικά στα πλοία μπορούσαμε να δούμε κάποιες λύσεις εφόσον ε, μπορούσαμε να ε, ανανεώσουμε τον εξοπλισμό με πολύ μεγάλο κέρδος ε, για την οικολογία για το περιβάλλον, να γίνει προσαρμογή των σκαφών ε, προς το πιο πράσινο και ίσως μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια μόχλευση του, των κονδυλίων χάρη στα ευρωομόλογα, τα ομόλογα έργου ε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ομόλογα έργου τα οποία ίσως δεν είναι τόσο απτά όσο το, το πραγματικό ζεστό χρήμα αλλά μπορεί να βοηθήσουν και να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι ένα μέσο πολύ σημαντικό για τις μεταφορές, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διαλειτουργικότητα και όπως είπε και η είναι δύο χωριστές οι εκθέσεις, ε, οι πρωτοβουλίες νομοθετικές. Χρειάζεται να μιλήσουμε ένα ψήφισμα για να προχωρήσουμε και στην Ολομέλεια. Εν γέννη, καλό σύνολο μέτρων χρήσιμο για τις πλωτές μεταφορές. Βαντάλεν. <clears throat> Eh, Ευχαριστώ. Αυτή η πρόταση παρουσιάζει δύο πτυχές. Πρώτον, μετά τη διαφωνία μεταξύ των ε, ε, αρμοδιοτήτων ε, ε, μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της περιοχής του Ρήνου, είναι καλό ότι μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία. Είναι όμως ένα απογοητευτικό πακέτο εξετάζοντας ε, το περιεχόμενο της Λευκής ε, Βίβλου, λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλή εξέλιξη των μέτρων για την εσωτερική ναυσιπλοεία, όμως όταν βλέπουμε τα 35 εκατομμύρια ευρώ, αυτό δεν είναι τίποτα πραγματικά. Ε, με τέτοιου είδους προϋπολογισμό είναι αδύνατον ε, την, ε, ε, τον, αφο, τον παροπλισμό αλλιευτικών σκαφών να τον επιτύχουμε. Μόνο, καλά, μόνο δηλώσεις καλών προθέσεων κάνουμε. Το Ταμείο Παροπλισμού. Είναι πολύ μικρό το ποσό ε, δεδομένων ε, των ηλικιωμένων στόλων που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη. Σίγουρα υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα σημεία στην πρόταση σε διάφορα σημεία, αλλά νομίζω ότι είναι απλώς ένα κείμενο το οποίο δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα την εσωτερική ναυσιπλοεία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στάινρουκ από την Επιτροπή απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ και για τη δική μου γνωμοδότηση από την Επιτροπή ε, Απασχόλησης. Ε, Καλώς ορίζω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στα θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας και την απασχόληση. Ε, έχουμε επικοινωνήσει και συνομιλήσει και με τις, τους εκπροσώπους των αλλιέων και με τους ε, εκπροσώπους ε, των εργαζομένων στον χώρο της αλίας και πιστεύουν όλοι, είναι σύμφωνοι ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δημορφωθεί δηλαδή, το Ταμείο έτσι ώστε να μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει. Έχει χαθεί πολλής χρόνος. Από το 1999 που δεν αξιοποιήθηκαν ή αξιοποιήθηκαν ε, ελλιπώς ε, τα κονδύλια αυτά. Ε, πρέπει να υπάρξει κάποια διατύπωση προς όφελος των δικαιούχων για τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους, ώστε να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην χρηματοδότηση αυτή. Για τον εξοπλισμό, για τον εξυγχρονισμό των στόλων θα πρέπει να υπάρξει αναφορά. Επίσης, και η δυνατότητα στην πρώιμη σταξιοδότηση, ε, χρηματοδότηση της ε, του τεχνολογικού εξυγχρονισμού και ε, βελτίωση της κατάρτισης των δεξιοτήτων του πληρώματος. Έτσι λοιπόν βελτίωση, ε, καλύτερος εξοπλισμός και μείωση του μεγέθους των σκαφών ή του δυναμικού είναι πολύ σημαντικές ε, διαστάσεις. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους. Ε, μιλήσαμε για μετακπαίδευση, κατάρτιση για να απτύξει άλλες δραστηριότητες. Μιλήσαμε για συνεργασία και με τους φορείς, τους εξοδοτικούς και με τα ταμεία ώστε να διαδίδουν ε, τις, τους ενδιαφερομένους τις πληροφορίες, να διαθέτουν τα φύλλα άδεια κτλ. Και για μένα επίσης είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων τυπικά στην ε, διαδικασία της διάθεσης των κονδυλίων, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά, καλύτερα από τον καθέναν τα προβλήματα, οι κοινωνικοί εταίροι. Έχω λοιπόν προτείνει κάποιες τροπολογίες. Στο άρθρο 1 ζητώ τα κράτη-μέλη να ε, αναπτύσσουν ε, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους τα μέτρα. Στην πρώτη παύλα ζητώ να σημειωθεί ενημέρωση για τις δυνατότητες είτε για ε, επανεκπαίδευση, επανακατάρτιση είτε για χρήση των κονδυλίων. Επίσης αναφέρω ρητά ε, ότι τα μέτρα αυτά προσφέρονται και στο πλήρωμα και αυτό αφορά όχι μόνο την κατάρτιση αλλά και τη δυνατότητα για πρώιμη σταξιοδότηση γιατί η Επιτροπή είχε αρχικά υπολογίσει μόνο τους ε, επιχειρηματίες αλλά νομίζω ότι πρέπει και το πλήρωμα να το βάλουμε μέσα στο σχέδιο αυτό. Επίσης ε, αναφέρομαι στα μέλη του πληρώματος, είτε πρόκειται για επιχειρηματίες, είτε πρόκειται για απασχολουμένους, ε, για μισθωτούς, ε, να έχουν μια καλύτερη ε, κατάρτιση εν γέννη. Έχω επίσης μια αναφορά στην ιδιαιτερότητα της ναυσιπλοεία εσωτερικών πλωτών οδών οργάνωση. Η Αρχική Ένωση Οργανώσεις ήταν πολύ ασαφής για μένα. Η κοινωνική εταίρη νομίζω είναι μια πολύ σαφής έννοια. Σε αυτούς κάνω εγώ ρητά αναφορά και πιστεύω ότι είναι και η καταλληλότερη ε, λύση. Επίσης μιλούμε για βελτίωση των συνθήκων εργασίας που θα πρέπει να συνοδεύονται από τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγιεινής στον χώρο εργασίας. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό εννοούσε και η Επιτροπή, αλλά δεν μου φάνηκε πολύ ξεκάθαρη η διατύπωσή της. Γι' αυτό και εγώ εδώ προτείνω μια πιο σαφή διατύπωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Φαντερέγγεν. Παρακαλώ λίγο σύντομα, γιατί πριν έρθει ο Λιθουανός υπουργό, θα ήθελα να, δώσω, να προλάβω να εξετάσω και την ε, έκθεση του κυρίου Λιμπεράτσκι. Ε, κύριε Φαντερέγγεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές ε, και της Επιτροπής Μεταφορών αλλά και της Επιτροπής ε, Απασχόλησης για την προετοιμασία της έκθεσης και του σχέδιου, του σχεδίου εκθέσεώς τους. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ουσία της έκθεσης που υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις ε, πτυχές που αφορούν ε, την ε, ικανότητα του στόλου. Θα ήθελα να πω ότι η πρόθεση της έκθεσης είναι να απελευθερώσει τα κονδύλια τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και υποστηρίζουμε την πρόταση του Κοινοβουλίου που κινείται προς την κατεύθυνση πράγματι της διεύρυνσης των δυνατοτήτων χρήσης αυτών των ε, κονδυλίων, ε, γιατί αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε μπορεί να υπάρξει τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα. Ε, ευχαρίστως λοιπόν να συζητήσουμε τις δυνατότητες της αξιοποίησης των κονδυλίων αυτών, να μην υπάρξουν επιπλέον ε, περιορισμοί και δυσκολίες για τη χρήση των κονδυλίων αυτών. Όσον αφορά την πρόταση τώρα για, τους, ε, για τις τεχνικές προδιαγραφές, και πάλι ε, συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με την άποψη του Κοινοβουλίου, Έχουμε κάποιες ε, ανησυχίες βέβαια σε σχέση με κάποιες υποχρεώσεις ε, υποβολής ε, εκθέσεων. Να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι στο πλαίσιο της ανακοίνωσης Ναϊάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη προβλέψει την έγκριση ενός σχεδίου ενός μιας εκθέσης πρόοδου Οπότε θεωρούμε ότι θα μπορούσατε τις πτυχές που συζητάτε να συμπεριλάβουμε, να τις συμπεριλάβουμε στις εκθέσεις πρόοδου αυτές. Και κάτι ακόμη, μία ακόμη πτυχή είναι ότι οι τεχνικές προδιαγραφές ε, για τα σκάφη εξελίσσονται συνεχώς και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα ήταν ε, σωστό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει ε, ε, εξουσίες εξουσιοδότησης ε, επειδή εξελίσσονται πάρα πολύ ακριβώς αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 15 ναι. Ιανουαρίου. Θα ψηφίσουμε 21 Ιανουαρίου. Ε, ξέρω ότι ο κύριος Γκρόσο τα σημειώνει όλα αυτά για την εισηγήτρια. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα που αφορά τις υπηρεσίες, τα οργανωμένα ταξίδια, ε, την έκθεση του κυρίου Λιμπεράτσκι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία ε, να μιλήσω, μια και είναι ο υπουργό εδώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ε, Ξέρει ότι υπάρχει μια οδηγία η οποία ε, υφίσταται από το 1999, εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, τεχνικές εξελίξεις, πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ. Βεβαίως εμείς θέλουμε όσο οι χρήστες μας ε, και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ε, να έχουν όσο γίνεται πιο ε, μεγάλη αξιοπιστία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αξιοπιστία. Θα πρέπει να ξέρει κανείς είτε ένας πελάτης, ένας χρήστης είτε αγοράσει εξατομικευμένο ταξίδι είτε οργανωμένο ταξίδι πρέπει να ξέρει ότι θα είναι ένα καλό ταξίδι, καλά οργανωμένο και αξιόπιστο, ότι θα υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία και με τους ε, διάφορους μεταφορείς, κυρίως αερομεταφορείς. Νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία, ε, εάν τα βάλουμε μαζί, τότε οπωσδήποτε ε, θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και ελπίζω ότι ε, θα είναι ευχαριστημένοι και οι χρήστες. Η κυρία Μέσνερ. Είσαι και η μόνη της εδώ. Ναι, ευχαριστώ. Όχι, είναι πολύ καλό που έχουμε αυτή την προσφορά γιατί είναι και σύμφωνη με τις με τα θέματα των δικαιωμάτων των ε, ε, επιβατών σε ταξίδια σε πακέτο, γιατί βέβαια και είναι διαφορετικές συνθήκες, άρα θέλουμε και την προστασία των ε, καταναλωτών και την αναλογία ως προς την τουριστική προσφορά, την υπηρεσία την τουριστική που προσφέρεται για να είναι το κριτήριο του τι σημαίνει προσφορά σε πακέτο αλλο η Προεδρία θα το καλύψει. Η Κομισιόν θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε τον ε, εισηγητή για την ε, έκθεσή του. Ε, θα θέλαμε να πούμε πάντως ότι έχουμε κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά τις τροπολογίες τις οποίες προτίθεται να προτείνει να επιστήσω την προσοχή σας ότι, πρέπει να ότι το προτινόμενο, ε, ε, το προτινόμενο επίπεδο ενερμόνησης είναι το χαμηλότερο δυνατό για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και σε σχέση με τον στόχο της πρότασης. Επίσης, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής έχουμε κάποιες, κάποιους ενδιασμούς ε, γιατί συστέλλεται το πεδίο εφαρμογής και επίσης ε, των ε, ε, ταξιδιωτικών διακανονισμών που ονομάζονται assisted travel arrangements, δηλαδή όχι ακριβώς πακέτο, αλλά παροχή εξατομικευμένων στοιχείων και εδώ νομίζουμε ότι συστέλλεται λίγο το πεδίο εφαρμογής. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε και κατά πόσον οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, υφίστανται αύξηση του άχθους. Πολλοί είναι οι πράκτορες ε, οι οποίοι αν δουν να εξελίσσεται προς αυτή την κατεύθυνση η κατάσταση και αν πρέπει να αναλάβουν την προστασία των καταναλωτών ε, θα αποφασίσουν ενδεχομένως να μην προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Όσον αφορά το θέμα ε, της ευθύνης είναι γεγονός ότι Εάν σε όλες τις χώρες ε, εισαχθεί η διπλή ευθύνη, τότε αυτό θα δημιουργήσει ενδεχομένως αύξηση ε, του κόστους των ταξιδιών. Επίσης, όσον αφορά κάποιες άλλες αλλαγές, όσον αφορά ε, την προστασία του καταναλωτή, όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων ε, ε, επισκοπού η Κομισιόν ε, δεν προτείνει ε, ε περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά τους μεμονωμένους ταξιδιώτες, τις μεμονωμένες ταξιδιωτικές ε, υπηρεσίες. Φοβόμαστε γενικά ότι κάποια από τα στοιχεία τα οποία προτείνονται εδώ μάλλον εμπίπτουν στην οδηγία για την προστασία των καταναλωτών και όχι στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Μετά από όλα αυτά βεβαίως που είπα, Πιστεύω ότι και μέσω των προτάσεων του εισηγητού μπορεί να βελτιωθεί ε, η ε, οδηγία. Οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε την συνεργασία ε, με, την Επιτροπή σας και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δεγκράντε, θέλετε να πείτε κάτι. Είναι εδώ ο υπουργό, περιμένει. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι οπωσδήποτε. Σύντομος να είστε πάντως. Sí, presidente, ε, ναι, ναι, έχουμε, έπρεπε να είχαμε χρόνο για τη συζήτηση, αλλά μας πήρε πολύ χρόνο ε, η ψηφοφορία και εδώ τώρα τι να σας πω, προχωράμε υπερβολικά γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πρόκειται για μια ιδιαίτερα ε, αναπόφευκτη θα πω πρόταση, γιατί πραγματικά άλλαξαν πάρα πολλά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ε, το ίντερνετ κτλ ε, και οι σχέσεις βέβαια και των καταναλωτών είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα όλα αυτά. Το είδαμε και με τα δικαιώματα των, ε, ε, το θέμα των δικαιωμάτων των ε, ταξιδιωτών. Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφάνεια. Δεν έχουμε δει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Βλέπουμε επίσης ε, να υπάρχει κάποια αντιπαράθεση ανάμεσα στον πραγματικό πάροχο της υπηρεσίας και αυτόν που ο καταναλωτής, ο χρήστης θεωρεί πάροχο της ε, ε, υπηρεσίας, διοργανωτή δηλαδή και μεσολαβητή. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν πλέον ξεπεραστεί και αυτά να τα διαγράψουμε. Ε, θα ε, έχουμε βεβαίως τροπολογίες προς, για να καλυφθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, η πρόταση αυτή θα πρέπει να γίνει όσο γίνεται σαφέστερη. Ε, οι ορισμοί, κυρίως ποιες είναι οι υπηρεσίες, ε, ποια είναι οργανωμένα ταξίδια, ποια είναι μεμονωμένα ταξίδια. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Το θέμα της ευθύνης επίσης είναι ε, απαραίτητο να ε, αντιμετωπιστεί, όπως άλλωστε το κάνει ο εισηγητής, έτσι ώστε να υπάρχει συνολική ευθύνη και από τον πολιτή της υπηρεσίας και από τον διοργανωτή. Επίσης, σε περιπτώσεις ε, λάθους ε, θα πρέπει να αναγνωρίζεται η συνολική ευθύνη. Δεν μπορεί ε, ο καταναλωτής να ψάχνει μόνος του και να βρει ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν σεβάστηκε τον ρόλο του. Είναι νέες οι σχέσεις οι οποίες προκύπτουν από, τη χρήση του ίντερνετ και θα πρέπει ο καταναλωτής να ξέρει ακριβώς με, ποιον έχει να κάνει, με ποιον υπογράφει τη σύμβαση, ποιος είναι υπεύθυνο και ποιος θα έχει τελικά την ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος όταν έχει αγοράσει ο καταναλωτής ένα οργανωμένο ταξίδι. Πρόεδρος, 18 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα, 16.00 δηλαδή, Ξέρω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το ε, ωράριο τέλο πάντων και τις προθεσμίες της ε, ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαστε όλοι πάρα πολύ σύντομοι. Το επόμενο θέμα στη ημερήσια διάταξη είναι η ε, παρουσίαση της, ε, της τελικής εισήγησης του Λιθιανού Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και πάλι εδώ αυτή τη φορά στο τέλος της ε, προεδρίας μας για να σας μιλήσω για την πρόοδο που επιτύχαμε τους τελευταίους έξι μήνες ως Λιθουανική Προεδρία. Όταν ήρθα τον Ιούλιο σας παρουσίασα το πρόγραμμα της Προεδρίας μας για το δεύτερο ήμιση της χρονιάς αυτής και σας είχα υποσχεθεί ότι η Λιθουανική Προεδρία θα ε, εξασφαλίσει τη συνέχεια, ε, τη συνέχιση της νομοθεσίας για τα διάφορα πακέτα και ότι θα συνεισφέρει στην, αξιόπιστη, στην δημιουργία μιας αξιόπιστης και ανοιχτής Ευρώπης. Όταν σας παρουσίασα το πρόγραμμά μας τον Ιούνιο, σας είχα πει επίσης ότι προσπαθώντας να επιτύχω αυτούς τους στόχους στον τομέα των μεταφορών, η Λιθουανία θα επιμείνει ε, στις τεχνολογικές εξελίξεις, ε, στις περιβαλλοντικώς φιλικές ε, μεταφορές, Επίσης, σας είχα μιλήσει για την ασφάλεια των οχημάτων και τη σχέση μεταξύ ε, των ε, δικτύων μεταφορών ε, που συνδέουν την Ευρώπη με τρίτες χώρες. Πριν κάνω έναν απολογισμό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου ιδιαίτερω του συναδέλφους στο Συμβούλιο για την επικοδομητική συνεργασία. Επίσης, ε, Brian, ε, είμαι και σε σένα πολύ ευγνώμων και στην Επιτροπή σας ε, για την επικοδομητική και αμοιβαία εποφελή εργασία, συνεργασία συγγνώμη, από την αρχή της Προεδρίας μας για μένα ήταν, ε, μια, ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα ε, σοφής πολιτικής ηγεσία. Θυμάμαι πολλούς εισηγητές με τους οποίους ε, συνεργάστηκα κατά τους τελευταίους έξι μήνες να ευχαριστήσω την κυρία Σενάλοβα, τον κύριο Φενκούν, ε, τον κύριο Χιστέλου, τον κύριο Ρικέ και την κυρία Ντεβεράκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους σκιώδεις εισηγητές και βεβαίως εσάς κυρίως κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω ε, από την κοινή προσέγγιση για την ε, οδηγία εναλλακτική υποδομής καυσίμων που ενέκρινε στις 5 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο Μεταφορών. Όπως γνωρίζετε, η οδηγία αυτή θέλει να ε, δημιουργήσει ανεξαρτησία από το ε, πετρέλαιο, ε, ένα καθαρότερο περιβάλλον και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να καταλήξουμε στη συμφωνία. Ήταν και άλλωστε μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας και πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μια βάση για ένα σύστημα μεταφορών αποτελεσματικό και αηφόρο. Συνεχίσαμε βέβαια τις προσπάθειές μας για να φτάσουμε σε μια, σε μια τελική ε, συμφωνία. Σήμερα έγινε η πρώτη συζήτηση με τον κύριο ε, Κάρλο Φιντάντσα, που είναι ο εισηγητής. Ε, συζητήσαμε μαζί του, είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας και νομίζω ότι τον Ιανουάριο του 2014, όταν θα ξαναρχίσουν οι εργασίε μα, θα υπάρχει μια πολύ καλή βάση για τη συνέχιση των συνομιλιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια για, το να, επιτύχουμε ε, στη, Συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για τον κανονισμό ε, GNSS, ε, δηλαδή τις δορυφορικές υπηρεσίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων μόλις ενέκρινε κοινή προσέγγιση για την οδηγία ε, που θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θα δώσει μια βάση για αποτελεσματικό ε, χωροταξικό σχεδιασμό στη θάλασσα, όπως για παράδειγμα την ε, μεταφορά ενέργειας από υπεράκτιες πλατφόρμες και τον τουρισμό. Νομίζω λοιπόν ότι στέλνουμε ένα καλό μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή ότι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να μπει σε διαπραγματεύσεις. Χαίρομαι που στον τομέα ε, των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου καταλήξαμε σε κοινή προσέγγιση για την αναθεώρηση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Είναι ένα τμήμα ε, των τεσσάρων ε, πακέτων για τους σιδηροδρόμους, του τέταρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους, συγγνώμη. Και σας παρουσιάσαμε επίσης σε μια έκθεση προόδου για τον κανονισμό ε, λειτουργίας ε, του οργανισμού ε, σιδηροδρομικών μεταφορών. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη ε, προεδρία θα συνεχιστεί η συζήτηση για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο θέμα των οδικών μεταφορών και του πόσο ε, καλή, καλή είναι οι οδικοί μας άξονες. Ε, είχαμε πει ότι θα θέλαμε να κάνουμε δοκιμές, ε, να υπάρχουν οδικές επιθεωρήσεις των οχημάτων, επιθεώρηση των εγγράφων, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να αυξηθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας στους δρόμους της Ευρώπης. Δεν ήταν εύκολες οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Είμαι πολύ ευγνώμονες, ε, είμαι ευγνώμονες ε, κυρίως εσένα Μπράιαν, ε, γιατί είχατε πάντοτε μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση προς το Συμβούλιο. Η Λιθουανία προσπάθησε πάρα πολύ για να υπάρξει πρόοδο σε σχέση με τις προτάσεις ε, για τα δικαιώματα των επιβατών, όπως για παράδειγμα καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη αποζημίωση για καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις ε, ή σε περίπτωση άρνηση επιβίβασης ε, σε ένα επιβάτη. Θα θυμάστε ότι αρχικά ο στόχος μας ήταν να συμφωνήσουμε για την κοινή προσέγγιση στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, όμως έπρεπε να αποδεχθούμε ότι το Συμβούλιο χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, χρειάζεται χρόνο να αποφασίσει νομικές πτυχές, όπως για παράδειγμα συμμόρφωση με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, όπως επίσης και τη συμμόρφωση των τρίτων χωρών. Η πρόταση αυτή έχει μεγάλη πολιτική σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μεριμνά για την προστασία των ε, επιβατών ε, των ε, αεροπλάνων και πρέπει να μην μας διαφεύγει ότι θα έχει πολύ σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε αεροπορικές εταιρείες αυτή η πρόταση. Επομένως πρέπει από την αρχή να τα κάνουμε όλα πολύ σωστά Έχουμε υποβάλει μία ε, περιεκτική έκθεση προόδου στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και θα συνεχίσουν οι συζητήσει σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Ω προ το θέμα τώρα των εναερίων μεταφορών, ε, θα ήθελα επίση να αναφερθώ σε μία συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία. Είμαι πολύ ικανοποιημένο για την έκβαση, γιατί έτσι βελτιώνεται η ασφάλεια των πτήσεων. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κριστίν Βεράκ, την εισηγήτριά μας και τους σκιώδεις εισηγητές, την εισηγήτριά σας τους ε, σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία. Επίσης, να επισημάνω το εξής ότι η διαδικασία διαβούλευσης έχει δρομολογηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν τω όμως το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει σε κοινή προσέγγιση ε, για την κοινοπραξία. Σίγουρα βέβαια θα ε, έρθουμε σε επαφή πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ε, συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο ε, αναμένεται για το θέμα της συγχωρήπανσης. Ε, έχουμε ήδη ένα έγγραφο με συμβαστικές προτάσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συνεχίσει η Ελληνική Προεδρία και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος ε, της κοινοβουλευτικής ε, θητείας. Ω προ το θέμα των θαλασσίων μεταφορών, έχουμε κοινή προσέγγιση για τον κανονισμό χρηματοδότηση ε, των δραστηριοτήτων τη Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Το, η συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο ήταν πολύ θετική, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα συμφωνία Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, τον Keith Taylor, όπως επίσης και εσάς για τη δική σας συνεισφορά, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στη συμφωνία σε αυτό το ευαίσθητο θέμα πολύ σύντομα. Θα ήθελα, επί τη ευκαιρία κύριε Πρόεδρε, να αφαιρθώ σε ορισμένα σημαντικά, σημαντικές εκδηλώσεις που οργάνωσε η Λιθουανική Προεδρία. Υπήρξε άτυπο Συμβούλιο Μεταφορών που έλαβε χώρα στο Βίλνιους στις 16 Σεπτεμβρίου. Τίτλος ήταν «Ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, μελλοντικό όραμα». Συζητήσαμε την πρόοδο, προ... την πρόοδο μας σε σχέση με το θέμα αυτό και συζητήσαμε για τις μελλοντικέ μας δράσεις οι Υπουργοί Μεταφορών, ε, Ευρωβουλευτές, ε, εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών ε, και πάροχοι υπηρεσιών αεροπλοείας συμμετείχαν στις συζητήσεις και επεσήμαναν την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας εναρμόνισης διαχείρισης της αναέρειας κυκλοφορίας οι στόχοι παραμένουν ίδιοι. Η ψηλότερη ασφάλεια στις πτήσεις, μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερη ασφάλεια του εναέριου χώρου, χαμηλότερο κόστος και μετριασμός, αν είναι δυνατόν, της ε, μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα αεροσκάφη, της μόλυνσης του ατμοσφαιρικού αέρα συγκεκριμένα. Επίσης έγινε μια συζήτηση με τους Υπουργούς Μεταφορών ε, ε, στο πλαίσιο της Ανατολικής ε, Γειτονίας τον Οκτώβριο στο Λουξεμβούργο. Οι Υπουργοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους για μια κοινή δήλωση για τη μελλοντική συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Επίσης εγκρίναμε ένα δίκτυο ε, μεταφορών ε, και συνεργασία με τις χώρες ανατολικής γειτονίας. Το δίκτυο αυτό συνεργασίας θα αποτελέσει τμήμα των μακροπρόθεσμων συνεπών πολιτικών μας ε, προς τους φίλους μας στην Ανατολική Ευρώπη. Με έξι χώρες εταίρους κυρίως ε, είχαμε επαφές, ε, γιατί θα υπάρξουν συγκεκριμένα προγράμματα με τις χώρες αυτές, ε, με χρηματοδότηση από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μάλιστα θέλαμε να συμπεριλάβουμε την προσπάθεια αυτή ε, στον κανονισμό κατευθυντηρίων γραμμών ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, η σύνοδος για την, στην Ανατολική Γειτονία που έγινε στο Βίλνιους στις 25 Νοεμβρίου τόνισε ότι ο τομέας εναέριας ε, κυκλοφορίας είναι ένα σημαντικό τμήμα της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των ανατολικών εταίρων μας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία του Συμβουλίου αποτέλεσε ε, μια νέα πρόκληση για μας, ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των φακέλων που είχαμε να εξετάσουμε όμως ε, θελήσαμε να ανταπεξέλθουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τομέα των μεταφορών και μπορώ να σας πω σήμερα ότι η Λιθουανία έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ε, για να υπάρξει γρήγορη πρόοδος ε, σε επίκαιρα θέματα και προκειμένου να διατηρήσει ή να εξασφαλίσει ευρεία συνένεση. Να ευχαριστήσω μία ακόμη φορά την Επιτροπή σας και εσένα προσωπικά, Brian, για την επικοδομητική πολύτιμη συνεργασία σου. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιητική έκφαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαρίστω να απαντήσω ερωτήσεις ε, για τα, ε, για τα μέλη της Επιτροπής σας. Κύριε Γκρός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους συνεργάτες σας προσπαθούν πάντα σε συνθήκες, όχι πάντα ευχερείς να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Η έκθεση του Βεγάκη για μας, ήταν για μας ένα πολύ θετικό μήνυμα για ένα πολύ απλό λόγο, διότι είχαμε την εντύπωση ε, με την έκθεση αυτή, αλλά λάβαμε και την επικύρωση αυτής της εντύπωσης εν τέλει, ότι μπορεί το Συμβούλιο όχι απλώς, το, κοινοβου... το Συμβούλιο να παραγνωρίζει το, το Κοινοβούλιο, αλλά και να υποτιμά το ρόλο του. Έχουμε λοιπόν ε, να κάνουμε με ένα ζήτημα το οποίο αφορά όχι μόνο εσάς ως Προεδρία αλλά γενικότερα το Συμβούλιο. Την εντύπωση δηλαδή ότι το Συμβούλιο κινείται πολύ αργά σε ορισμένα θέματα και ότι ε, πολύ συχνά μας λέει ότι συμμερίζεται τους στόχους μας με ωραία λόγια κτλ. Αλλά δεν ακολουθούν τα ωραία αυτά λόγια και τα αντίστοιχα έργα. Όλο αυτό το πακέτο παραδείγματι των προτάσεων για τις ενέργειες μεταφορές με τους τρεις φακέλους, τα, τρία νομοθετήματα που εγκρίθηκαν και για τα οποία δεν έχουμε καμία πρόοδο εκτός από ένα. Ε, η προοπτική να έχουμε τους ενιαίους ουρανούς, ενός ευρωπαϊκούς ουρανούς, δεν φαίνεται τόσο κοντά. Ε, οι στόχοι που υποστηρίζουμε εμείς είναι και πιο οικολογικοί και πιο εύχρηστοι και πιο ασφαλείς. Ε, και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε και γι' αυτό άλλωστε και θα καταθέσει φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέες προτάσεις που θα απασχολήσουν και πάλι το Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει για τους συντηροδρόμους θα ήθελα να σας πω το εξής ξεκινήσατε σε, τις, εργασίες σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το τεχνικό, στον τεχνικό τομέα, γιατί η διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητο στοιχείο των σιδηροδρόμων. Διαφορετικά δεν μπορούμε ποτέ να μιλούμε για εναρμόνιση στους σιδηροδρόμους. Είναι πολύ, πολύ έντονες οι τεχνικές διαφορές. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πακέτο, το οποίο πρέπει να μείνει πακέτο, όπως και να έχει, έστω και αν ξεκινήσετε από ένα κομμάτι του. Και βεβαίως το πακέτο αυτό έρχεται και λαμβάνει πολύ μεγάλη σημασία το ζήτημα των δικαιωμάτων των επιβατών, των καταναλωτών και σε αυτό ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας, τη βοήθειά σας ώστε να προχωρήσει το θέμα αυτό και να ευοδοθεί. Για τους ελέγχους ε, και τους, τους δρόμους ήταν πολύ δύσκολο θέμα. Ξέρω ότι νέρωσαν πολύ το κρασί τους ορισμένοι συνάδελφοι και τους ε, ευχαριστώ επ' ευκαιρία. Ήταν πολύ περιορισμένο το περιθώριο ε, κινητικότητας του Συμβουλίου, του Συμβουλίου σε σχέση με αυτά που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο και ε, με όλες τις ε, αντιφάσεις και τις θέσεις που είχαν εκφράσει στη συζήτηση. Πάντως πιστεύουμε ότι μπορεί να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν για τις προσπάθειές σας, αλλά να μεταφέρετε παρακαλώ και το μήνυμα προς το Συμβούλιο ότι για τα επόμενα σημαντικά θέματα πρέπει να ολοκληρωθούν και στην τρέχουσα μάλιστα θητεία κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Οι καθυστερήσεις δεν εξυπηρετούν το συμφέρον ούτε τη Ευρώπη ούτε των πολιτών μας και σε αυτό περιμένουμε, αναμένουμε την πλήρη υποστήριξή σας. Κύριος Αλκαντράου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Υπουργό για την τοποθέτησή του, για την ομιλία. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο το έργο της Προεδρίας, τώρα που ολοκληρώνεται νομίζω μπορούμε να το πούμε. Ε, Πάντως θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκρός, ε, ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα, έχουμε σε μερικούς μήνες ευρωεκλογέ. το κοινοβούλιο λίγο πολύ θα αρχίσει να αδρανεί και ε, έχετε τώρα τη χρυσή ευκαιρία να ολοκληρώσετε, να κλείσετε κάποια σημαντικά θέματα. Τώρα όμως. Γι' αυτό και ε, λυπούμαστε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι σε ορισμένα θέματα δεν μπορέσατε να ε, κλείσετε, να καταλήξετε συμφωνίες. Η ΕΜΣΑ, το πακέτο για του σιδηροδρόμους, είναι παραδείγματι που ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία και πιστεύω ότι θα, μπορέσα, θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις. Τα επτά διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών επίσης που είχαν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ή μάλλον του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και δεν έχουν προχωρήσει καθόλου εντωμεταξύ. Στο τελευταίο συμβούλιο, συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας ε, διαπιστώσαμε ότι πολλές ε, εκθέσεις προόδου ακούσαμε να παρουσιάζονται, αλλά πρόοδο δεν είδαμε. Και ένα σημαντικό πακέτο των ενέργων μεταφορών και των σιδηροδρόμων που με πολύ κόπο που εξεργαστήκαμε, πολύ εντατική δουλειά. Ε, όπως και πολλά άλλα βέβαια θέματα πρέπει να προχωρήσουν. Έχετε κάθε συμφέρον να προωθήσετε τις μεταφορές στην Ευρώπη, την πολιτική των μεταφορών. Και ξέρω ότι είναι συλλογικό όργανο το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι εδώ και χρόνια ε, καρκινοβατεί στις εργασίες τους τομείς αυτούς και ξέρουμε επίσης στον χώρο των μεταφορών πολύ ε, δίνουν την εντύπωση ότι οι πολύ λίγοι αντίθετα είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται με ευρωπαϊκή προοπτική. Αλλά δεν κάνει κακό να υπενθυμίζουμε, να κάνουμε μια υπόμνηση ε, στα θέματα αυτά και να τσιγκλάμε λίγο. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε τους ομάδες μου. Ευχαριστούμε για όσα κάνατε. Και τώρα, που ξέρετε και τι είναι να έχει κανείς ε, αναλάβει η Προεδρία, και με την ελπίδα ότι θα σας ε, έχουν κοπεί τελείως τα φτερά και ότι θα μπορέσετε να εργαστείτε καλά στους επόμενους μήνες και να συνεργαστείτε με την προσεχή Προεδρία. Ελπίζουμε ότι θα ε, ευοδοθούν αυτοί οι φάκελοι. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Υπουργό για την ομιλία λήξης της Προεδρίας. Δεν έχω να πω και πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που είπαν οι δύο προλαλήσαντες. Θα το έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι και εσείς. Ότι εμείς εδώ ως βουλευτές προερχόμενοι από όλα τα κράτη-μέλη και από κόμματα που έχουν κυβέρνηση στα κράτη-μέλη βρισκόμαστε πολύ συχνά σε αντίθεση, σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις αυτές, ακόμη και αν είναι από τα δικά μας κόμματα. Και προσπαθούμε να κάνουμε καλά νομοθετήματα, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην Προεδρία του Συμβουλίου. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει, ναι, έστω να κάνει και το ρόλο του θηριοδαμαστεί ώρες ώρες για τα κράτη-μέλη, αλλά πάντως πρέπει να φέρνει αποτελέσματα. Ε, ήταν αυτή η πρώτη σας ε, προεδρία, μεγάλες οι προκλήσεις που είχατε να αντιμετωπίσετε. Είχατε ένα τεράστιο όγκο νομοθετημάτων ε, να διεκπαιρεώσετε σε αυτό το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής θητείας, θέματα τα οποία έπρεπε να προχωρήσουν πριν σταματήσουν οι εργασίες. Αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα ο χώρος των μεταφορών στην Ευρώπη για τους πολίτες, για τις ευρωπαϊκές μεταφορές είναι ο στόχος για τον οποίο εργαζόμαστε όλοι. Εγώ δεν έχω λάβει μέρο σε τόσους ε, πολλούς τριμερεί διαλόγους από το που έχω αναλάβει την θέση του συντονιστή. Έχω μια κάπω γενικότερη επισκόπηση, αλλά στο θέμα του roadworthiness, ε, δηλαδή της αξιολόγησης ε, καταλληλότητας για τις μεταφορές, για τους οδικές μεταφορές ενός οχήματος, όπως τακταίο και συναφείς οργανισμοί, νομίζω ότι Θέλουμε βεβαίω την αναρμόνιση για την ασφάλεια των δρόμων. Δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τι πρόοδου. Για του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ξέρω ότι είναι πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει μένα, αλλά κανένα δεν έχει αναλογιστεί ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και ώρα να εφαρμόσει τα όσα έχει υπογράψει. Αυτό ανέξαρτος του ποια είναι η, χώρα που έχει την Προεδρία, οπωσδήποτε πρέπει κανείς να προσπαθήσει να φέρει κάποια κινητικότητα. Ε, με τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς είμαστε και ανυπόμονοι, βρίσκοντας στο Κοινοβούλιο και πολλές φορές εξοργιζόμαστε με τα κράτη-μέλη και βέβαια αυτά τα εισπράττει η Προεδρία. Ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα καλύφθηκαν ήδη και το Linking Europe Facility ε, από το 2009 που είμαι εγώ στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι δεν έχουν συναντήσει άλλα θέματα, άλλες προτάσεις πολιτικής ε, τέτοια υποστήριξη όσο το να συνδεθεί η Ευρώπη ε, και να εκφραστεί μέσα σε ένα χάρτη το σύστημα των μεταφορών της αντίστοιχο με έναν χάρτη του μετρό. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά. Είχαμε προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες φαινόντουσαν πολύ καλές επί παραδείγματι η οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων. Ένα θέμα δύσκολο. Όπου ακόμα και το ζήτημα της γλώσσας ε, αποτέλεσε πρόβλημα και δεν μπόρεσε να πλησιάσει, να προσεγγίσει τις θέσεις μας η διαπραγματεύτρια στο Συμβούλιο. Ε, η, ο κανονισ... η χωροταξία, η θαλάσσια χωροταξία στην οποία είμαι εγώ αρμόδια είναι ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, το έχουμε συζητήσει. Και ξέρω ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία στο Συμβούλιο, αλλά πρέπει πια να προχωρήσουμε. Αν είναι έτοιμο και το Συμβούλιο, φαντάζομαι ότι η Επιτροπή είναι ήδη έτοιμη να προχωρήσουμε. Έστω και αν κάποια πράγματα μένουν ε, ελλειπή σε σχέση με αυτά θα ήθελα εγώ. Επίσης ε, η υποδομή για εναλλακτικέ μορφές ενέργειας ξεκινάει τώρα με ένα πρώτο τριμερή διάλογο. Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν προκαταβολικά κάποια σημεία για να μην χρειαστεί η διαπραγμάτευση να επεκταθεί στα πάντα. Ε, σε αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή και πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Σενάλοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Όταν η Λιθουανική Προεδρία ανέφερε και τα στοιχεία τα οποία ε, είχε σκοπό να θίξει ε, είχε αναφερθεί ε, και σε ένα πακέτο για τους ελέγχους τους αυτοκινητοδρόμους. Ήμουν εγώ η συγγήτρια μάλιστα. Προσπαθήσαμε έτσι ώστε η Πολυθουανική Προεδρία να επιτύχουμε κάποια αποτελέσματα. Κάναμε κάποιες τεχνικές συναντήσεις και ε, επιτέλους ε, τώρα φτάνουμε και σε μια πάρα πολύ δύσκολη συμβαστική λύση, την οποία όμως επιτύχαμε. Έστω και αν Λυπούμε γιατί το Συμβούλιο υπό την λιθουανική ηγεσία ε, δεν έδειξε μεγαλύτερη φιλοδοξία γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ε, αυτή η νομοθεσία είναι σημαντική και τα μάλλα μπορεί να συμβάλλει ε, στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων. Εν πάση περιπτώσει Είμαι και λίγο απογοητευμένη και σε ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται πάλι με την οδική ασφάλεια. Αυτή η έλλειψη αναλογίας, αυτή η δυσαναλογία σε σχέση με το πόσο μακριά καταφέραμε να πάμε με την, ε, το, κοινοβούλιο δηλαδή όσον αφορά την ηλεκτρονική κλίση e-call και μέχρι που έχει φτάσει το Συμβούλιο. Ε, τώρα δηλαδή αρχίζει να δουλεύει για το θέμα αυτό το Συμβούλιο. Όταν λοιπόν θα δώσετε την προεδρία στη, στους Έλληνες συναδέλφους σας, ε, μήπως μπορείτε να τους πείτε να πιέσουν, γιατί επίγουν τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριο Κούν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω όμως κάποια ε, αυροφροσύνη στην ε, Λιθουανική Προεδρία για την πρόοδο, για την όποια πρόοδο κατάφερε σε αυτούς τους φακέλους. Έτσι είστε τόσο μικρή ε, χώρα όσο το Μεκλεμβούργο, Άνω Πομερανία, που είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο το ότι καταφέρατε αυτό και οφείλουμε συγχαρητήρια στον Υπουργό, ήταν στο High Level Group, στο Συμβούλιο, ένας από εκείνους οι οποίοι πράγματι επισήλθαν στις λεπτομέρειες και συζητήθηκε ένα παράρτημα 80 σελίδων με ελάχιστες προδιαγραφές εντός εισαγωγικών που συμφωνήθηκαν για την επιθεώρηση οχημάτων με κινητήρα ε, σειρώμενων, ρημουλκών, ρημουλκούμενων ε, και τέτοιων ε, οχημάτων για μια μακρύτερη στο περίοδο για το 2000, έως το 2022 ε, και νομίζω ότι όπως και να έχει αυτό το φάκελο για, τον, για την καταλληλότητα, για το οδικό δίκτυο των οχημάτων και το ανέφερε η νωρίτερα, μέσα στην Ευρώπη πρέπει να έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές ορατές και αυτό πρέπει να το πούμε, οι οποίες μάλιστα εφόσον τηρούνται και στο συνεργείο και στην επιθεώρηση τεχνική, τότε βελτιώνουμε ασφαλώς την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα για τα κράτη που είναι κράτη ε, διέλευσης όπως η Γερμανία. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό Και ξέρετε ότι παλιά είχαμε με, τους, με τις κάτω χώρες την πρωτοπορία στον τομέα αυτόν, αλλά τώρα με τη διεύρυνση προς Ανατολάς τα πράγματα αλλάζουν, υπάρχουν πολύ διαφορετικές προδιαγραφές και πρέπει να υπάρχει η ετήσια οπωσδήποτε επιθεώρηση καταλληλότητας, τεχνική επιθεώρηση για τα οχήματα και τα ιδιωτική χρήσεως βεβαίως. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον κάθε πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά βεβαίω. Αλλά ήθελα να πω ότι από δική σα πλευρά τουλάχιστον ήταν αξιόλογο, πολύ αξιόλογο αυτό που κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ε, ευχαριστώ πολύ για τις καλές σας ιδέες. Μπορώ να σας πω ότι όποτε έρχομαι ότι ερχόμενος μάλλον εδώ, ε, δεν, ε, στην συνεδρία της σας, δεν περίμενα να μου δώσετε μετάλλιο, του αντίον μάλιστα. Ε, περίμενα ότι θα μου πείτε ότι θα έπρεπε να είχαμε δουλέψει πιο γρήγορα, ότι θα έπρεπε να είχαμε συζητήσει πιο πολλά θέματα, ότι θα έπρεπε να είχαμε επιτύχει περισσότερα αποτελέσματα. Ανοιχτά πάντως τώρα μπορώ να σας πω ότι οι ιδέες σας είναι απολύτως ορθές και αυτές αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για μένα ως Υπουργό. Θα συζητήσω όλα αυτά τα θέματα ε, με την Ελληνική Προεδρία και πιστεύω ότι ε, θα είναι εποφελές ε, ε, αυτό. Είχα παρουσιάσει τις ε, πρωτοβουλίες μας ε, λίγο ένα εξάμεινο πριν και νομίζω ότι πολλά πετύχαμε από αυτά τα οποία είχαμε θέσει ως αρχές αλλά βεβαίως ε, καμιά φορά ε, κανείς έχει πολλές επιθυμίες αλλά ε, του λείπουν οι δυνατότητες οι συγκεκριμένες για να επιτύχει κάποια πράγματα. Έρχονται εκλογές, το ξέρουμε εμείς, έχουμε Έχουμε πετύχει αρκετά. Ε, τώρα είναι η δικιά σας σειρά βέβαια να ε, εκτεθείτε στην ψήφο. Ελπίζω να έχετε καλή τύχη και στις εκλογές και μια και έρχονται Χριστούγεννα να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχές στο νέο έτος θα θέλαμε και εμείς να σας ευχηθούμε σε εσά και την οικογένειά σας και το, όλους τους ανθρώπους της ομάδας σας να σας ευχηθώ λέω καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Καλά Χριστούγεννα και ε, ευτυχές το νέο έτος. Ορίστε, σας έχω και ένα δωράκι. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σίμψον. That's my new, looks like my new tie. Yeah, yeah. Α, μάλλον ε, θα είναι η γραβάτα που θα λανσάρω τώρα, η καινούργια μου γραβάτα. Okay, folks, just to tell you now that... Λοιπόν, να σας πω από τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, Α, θέλεις κάτι? Ναι. Μια και είναι κάπως εξεχωριστή αυτή η μέρα και το έχω συζητήσει και με τους άλλους γεωδησίτες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στο να κάνουμε τις ψηφοφορίες με καλούς καταλόγους ψηφοφοριών. Ήταν πολύ σκληρή η δουλειά που έκανε η γραμματεία και όλοι οι άλλοι του προσωπικού μας που βοήθησαν και εκ μέρους και του συναδέλφου Αλκατράου αλλά και των λοιπόν νομίζω οφείλουμε να πούμε συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πραγματικά πολύ ειδικέ συνθήκες. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλο το προσωπικό, η βοηθή, ε, η βοηθή των βουλευτών, ε, η βοηθή εδώ, η γραμματεία, οι διερμηνείς, ε, όλοι βοήθησαν σήμερα έτσι ώστε αυτά τα τόσο τεχνικά ζητήματα να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε μέσα σε μία μέρα και Κοιτάξτε, βέβαια κουραστήκαμε. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι πρέπει να κοιμηθώ μια εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το αναγνωρίσατε. 9 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί θα ξανασυναντηθούμε. Να σας ευχηθώ πολύ καλά Χριστούγεννα, ευτυχέστατο το νέο έτος. Τις ίδιες ευχές ε, προς τους διερμήνες και τις οικογένειές τους ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. και μετά θα αρχίσει η τελική ευθεία βέβαια για το Κοινοβούλιο. Όλοι όσοι μας κοιτούν μέσω webcam, ε, γιατί τους λησμονούμε. Να τους ευχηθούμε λοιπόν όσους μας παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου. Ε, να, να τους ευχαριστήσουμε, να ελπίσουμε και να ευχηθούμε ότι και του χρόνου θα μας παρακολουθούν με την ίδια αδημονία ε, χρόνια πολλά και σε όλους. Τελείωσε η συνεδρίασή μας. Ευχαριστούμε πολύ.